Θα ψηφιστεί έκθεση του κύριου Μπέρμαν το μεσημέρι. Έχω μερικέ ανακοινώσει τώρα. Σύμφωνα με το άρθρο 216 παράγραφος 4 σας ενημερώνω ότι δεν έχει ζητήσει κανείς να ψηφιστεί το διορθωτικό που ανακοινώθηκε εχθές στις 5.30. Αυτά τα διορθωτικά λοιπόν θεωρούνται και Σε ό,τι αφορά τις συστάσεις απόφασης Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτού Εχτές αποφασίστηκε ότι δεν θα προβληθεί αντίρρηση ε, στις προϋποθέσεις δημοσίευσης ε, στην ε, ιστοσελίδα και στο διαδίκτυο για κάποια